Okay. Αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα, καλωσορίζω εδώ όλους τους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων σε αυτήν την διακοινοβουλευτική συνεδρίαση που οργανώνει η Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα τελευταία χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή μας, η Οικονομική Επιτροπή, θέλει να διασφαλίσει ότι οι μεταρρυθμίσεις της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και οι άλλες που έχουν να κάνουν με την μετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφύγης, συνοδεύονται από δημοκρατική λογοδοσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει πάντα τη συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, σας υπενθυμίζω ότι χωρίστε σε δύο τμήματα η σημερινή μας συνεδρίαση, ε, μια ώρα στο κάθε τμήμα. Στο πρώτο τμήμα θα ανταλλάξουμε απόψει όσον αφορά την φορολογία και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο εξή ερώτημα. Πώς και, τι ε, θα, και πώς θα έπρεπε να είναι ένα διεθνές φορολογικό σύστημα. Και το δεύτερο τμήμα θα ασχοληθεί με θέματα όπως είναι η διαφάνεια, η βιωσιμότητα και η περιβαλλοντική κοινωνική στόχη, όπως επίσης και η στόχοι διακυβέρνησης στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Επειδή είμαστε πάρα πολλοί, δεν θα μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο, οπότε θα φροντίσουμε, αν μη τι άλλο, όσο γίνεται ε, περισσότερα σώματα που εκπροσωπούνται εδώ κοινοβουλευτικά θα πάρουν το λόγο. Έτσι, δύο λεπτά θα έχει το λόγο ο καθένας για την κάθε του παρέμβαση. Ε, θα έχουμε δηλαδή 15 με 20 παρεμβάσεις το πολύ σε κάθε τιμή μας συζήτησης. Και ανάλογα με τις εξελίξεις της συζήτηση, τα χρονικά αυτά όρια θα προσαρμοστούν ανάλογα. Επίσης, υπάρχουν κάρτες για να ζητήσετε ε, χρόνο ομιλίας. Για να δω αν έχω εδώ. Είναι μία πράσινη, δεν την έχω εδώ πέρα μαζί μου, αλλά πρέπει να έχετε μπροστά σας ένα πράσινο χαρτί. Να, έτσι ακριβώς είναι αυτές οι κάρτες για χρόνο ομιλίας. Πρέπει να τις συμπληρώσετε λοιπόν. Αν θέλετε να πάρετε το λόγο και να τη δώσετε σας παρακαλώ στους κλητήρες. Έπειτα θα έχουμε τρεις εθνικούς βουλευτές και έναν ευρωβουλευτή που θα παίρνουν το λόγο και ούτω καθεξής. Τώρα και πάλι και αυτό το σύστημα μπορεί να χρειαστεί να προσαρμοστεί. Καλωσορίζω εδώ και δίνω και το λόγο στον Αντιπρόεδρο Μπόρις Λάλοβακ για να σας καλωσορίσει και αυτός εδώ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω κροατικά. Αξιότιμοι σας και συνάδελφοι, Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που σας καλωσορίζω εδώ σήμερα στις Βρυξέλλες εκ μέρους των ε, βουλευτών ε, και ανδρών και γυναικών της Κροατικής Βουλής και μου προσωπικά. Μετά από 30 χρόνια η Κροατική Δημοκρατία ε, έχει την χαρά και την τιμή να ασκεί την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι γιατί θα δώσουμε και εμείς τη δική μας συνεισφορά στα πλαίσια του νομοθετικού κύκλου σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Και μάλιστα από τη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Οικονομικών της Κρατικής Βουλής αλλά και ως πρώην Υπουργό Οικονομικών είμαι πεπισμένος ότι η σημερινή συζήτηση θα είναι πολύ επικοδομητική και θα μας δώσει έμπνευση για περαιτέρω εργασίες. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε το πρώτο τμήμα της συνεδρίασης που είναι αφιερωμένο στις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το διεθνές φορολογικό σύστημα. Η ψηφιοποίηση και η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει αυξήσει πάρα πολύ τη γεωγραφική κινητικότητα όσον αφορά την φορολογική βάση και οι πολυεθνικές έχουν να παίξουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο διεθνές εμπόριο. Πράγματι, οι προηγούμενες δεκαετίες τα συστήματα τα φορολογικά ήταν διαφορετικά. Για να ανταποκριθούμε λοιπόν στι διάφορε πιέσει, οι κυβερνήσει εργάζονται προκειμένου να μεταρρυθμίσουν τα φορολογικά του συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων όσον αφορά την εφαρμογή της ε, βάσης ε, διάβρωσης και της μεταφοράς ε, κερδών, τα σχέδια δηλαδή τα οποία εκπονούν η G20 και όσα. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχει εισάγει με τη στήριξη του Εθνικού Κοινοβουλίου νέα μέτρα. Οι φορολογικές αρχές επίσης προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το θέμα με συστάσεις αναχώρα με, για τις πολυεθνικές και για τους ενδιάμεσους οι οποίοι πρέπει πάντα να εντοπίζουν τα προγράμματά τους τα οποία χρησιμοποιούν επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια σημαντική πρόταση, μάλλον όχι μόνο μία, περισσότερες, προκειμένου να συγχρονίσει το σύστημα πληρωμή τη φορολογία από πλευρά των επιχειρήσεων ε, ακόμα και εκείνων που δεν βρίσκονται με φυσική παρουσία στην επικράτειά τους. Παράλληλα υπάρχουν συζητήσει ε, στο επίπεδο των G20 και του ΟΟΣΑ με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τα τέλη αυτής της χρονιάς. Το 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία ψήφισμα για την δίκαια φορολόγηση μέσα σε μια οικονομία που είναι ψηφιοποιημένη και παγκοσμιοποιημένη. Στο ψήφισμα αυτό, οι ευρωβουλευτέ εκφράζουν την ανησυχία του, λέγοντα ότι δεν υπάρχει κοινή προσέγγιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για τι ε, διαπραγματεύσει που λαμβάνουν χώρα σε διεθνέ επίπεδο και ζήτησε από την Επιτροπή και τι χώρε μέλη να αποφασίσουν για μια κοινή και φιλόδοξη θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει με μία φωνή και να αποτελέσει παράδειγμα ώστε η φορολόγηση να είναι δίκαια για όλους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το τόνισε αυτό ξανά και ξανά στη συζήτηση και εδώ θα υπενθυμίσω τρία κυρίω στοιχεία. Πρώτον, ότι δεν πρέπει να περιορίζουμε την ψηφιακή οικονομία και να δούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το διεθνές φορολογικό σύστημα που δεν οφείλεται μόνο στην ψηφιοποίηση της οικονομίας μας αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι η οικονομία μας ε, λειτουργεί μέσα σε όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να προχωρήσουν προς κάθε πλευρά. Έπειτα, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το θέμα της φυσικής παρουσίας μιας επιχειρήσης, δεν πρέπει να φορολογείται μόνο εφόσον έχει φυσική παρουσία σε μια χώρα, αλλά να τονίσουμε ότι το δίκτυο των έξω θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται με πολίτες, ε, με πελάτες και χρήστες, ακόμα και ψηφιακά. Και τρίτον, λέμε ότι σε σχέση με τον κανόνα εσόδων, το ελάχιστο επίπεδο φορολόγησης θα πρέπει να τεθεί για κάθε δικαιοδοσία όπου βρίσκονται πολυεθνικές, ώστε να υπάρχουν όλο και λιγότερες δυνατότητες για αυτές να προχωρούν σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο για να έχουμε μια, ε, ένα καλό και αποτελεσματικό σύστημα, γιατί πρέπει έτσι να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες και την αστάθεια. Ω Ευρωβουλευτέ, χρέο μα είναι να συνεχίσουμε να ελέγχουμε και να υποπτεύουμε την πρόοδο που γίνεται από τι κυβερνήσει μα επ' αυτού. Πρέπει να πιέσουμε τι κυβερνήσει μα για να διασφαλίσουν ότι οι μεγάλε πολυεθνικέ πληρώνουν το μερίδιο που πρέπει να πληρώνουν στη φορολογία αλλά πρέπει να βρεθούν και λύσεις έτσι ώστε οι, τα αποτελέσματα και οι αποφάσεις να είναι ισόρροπες και ισότιμες για όλους. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τον κύριο Τζεντιλόνη που είναι Επίτροπος για την Οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. στη συνέχεια τον ε, κύριο Πασκάλ Σενταμάς που είναι Διευθυντής για την Φορολογία στον ΟΣΑ, στη συνέχεια την κυρία Γκορτζάνα Πέρι, που είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών και Κεντρικού Προπολογισμού στο Κρατικό Κοινοβούλιο και τον κύριο Χάνης Μίχελμπαχ επίση, που είναι από το ΕΛΚΑ και συμμετέχει στην Επιτροπή Οικονομικών της Γερμανικής Bundesbank. Λοιπόν, πρέπει να απαντήσουμε στο εξή ερώτημα. Τι ρόλο πιστεύετε ότι πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ταπιστούν οι προκλήσεις από την φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να παίζει ηγετικό ρόλο στα πλαίσια του όσα σήμερα. Και τέλος, πώς να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες μέλη μπορούν να συμφωνήσουν ή όχι για μια φιλόδοξη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μεταρρύθμιση αυτή σε διεθνές επίπεδο. Ξεκινάει η συζήτηση λοιπόν και για πέντε λεπτά θα δώσω το λόγο στον Πάολο Τζεντιλόνι. Παρακαλώ. Uh, well, thank Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ επίκαιρο θέμα για τα κοινοβούλια. Το πιο επίκαιρο και το πιο σημαντικό για τα κοινοβούλια είναι η φορολόγηση. Αν εξετάσουμε τα τρία βασικά θέματα που συζητούνται, βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κάποια πρόοδο. Αλλά έχουμε τρία βασικά θέματα μπροστά μας. Το πρώτο, χρειάζεται να συνεχίσουμε την καταπολέμηση της φόρα αποφυγής και των φορολογικών ε, παραδείσων. Σήμερα σωστά το Συμβούλιο επικαιροποίησε τον κατάλογο των νομοθεσιών των ενόμων τάξεων που δεν συμμορφώνονται, το μαύρο κατάλογο, τη μαύρη λίστα, Προσθέσαμε τέσσερις νέες χώρες και επικράτειες. δεύτερο να δούμε πώς αλλάζουν τα φορολογικά μας συστήματα ανάλογα με την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας με το Πράσινο Σύμφωνο. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας, να αλλάξουμε την οδηγία για τη χρήση ενέργειας και συνεχίζονται οι εργασίες όσον αφορά την προσαρμογή, τη φορολογική προσαρμογή στα σύνορα όσον αφορά τη διαρροή άνθρακα. Θέλουμε να προστατεύσουμε τις διαρροές, να προστατευτούμε από τις διαρροές άνθρακα και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις κατά τις οποίες εξωτερικές οικονομίες μπορεί να έχουν λιγότερο φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους από ό,τι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν θέλουμε να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους, πρέπει να ετοιμάσουμε μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε τις σχετικέ αρνητικές συνέπειες. Τρίτο θέμα. Τα παγκόσμια θέματα. Οι προτάσει του ΩΣΑ. Θέματα που θα συζητηθούν αυτό το Σαββατοκυριακό. Στο ΡΙΑΝΤ. Στη σύνοδο των G20, των Υπουργών Οικονομικών των G20 Εκεί θα εκπροσωπήσω εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτό το τομέα πρέπει να πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα αυτά που είπε η κυρία Πρόεδρος για τις αρχές που ακολουθούμε. Έχουμε μία θετική συμφωνία τεχνικής φύσεως που ενετάχθη στο πλαίσιο του ΟΣΑ τέλος Ιανουαρίου στην τεχνική φύσεω συμφωνία υπάρχει όμως διαφοροποίηση των θέσεων ενός κράτους μέλους, των Ηνωμένων Πολιτειών, πολύ σημαντική χώρα, ζητά η χώρα αυτή να ακολουθηθεί, να εξεταστεί και διαφορετικό ενδεχόμενο. Αυτό που η Αμερικανική κυβέρνηση αποκαλεί ας μηχανισμός το ασφαλούς λιμένος. Δύσκολο να μεταφραστεί αυτός ο όρος παρά να το πούμε ερεσιμότητα, επιλεξιμότητα. Να επιτρέπουμε στις εταιρείε να επιλέγουν για τη φορολογία τους που θα καταβάλουν το φόρο. Αυτό καθιστά μια παγκόσμια εμβέλεια λύση σχετικά πίθανη, αυτή η απέτηση τον είπα. Έχουμε πολλές δυνατότητες για να συνεχίσουμε τη διαδικασία στο Ριάντ ίσως δεν κάνουμε το αποφασιστικό βήμα, αλλά ένα απλό βήμα προόδου, καλό βήμα, να εξακολουθούν να σκούνται πιέσει και να καταφέρουμε τον επόμενο Ιούλιο να βρούμε μια λύση. Είναι κρίσιμη σημασία να βρούμε λύση. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι χωρίς μια παγκόσμια λύση και με κάποια ευρωπαϊκά κράτη-μέλη να έχουν εθνική νομοθεσία που ακολουθούν σε αυτά τα θέματα και με το κίνδυνο αντιπίνων από πλευράς κυβερνήσεως των ΗΠΑ όσον αφορά τα εμπορικά ζητήματα μπαίνουμε σε πολύ επικίνδυνες ε, καταστάσεις προς αντιμετώπιση. Πρέπει να πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειες για μια παγκόσμια λύση. Ψηφιακοί γίγαντες επίσης υποστηρίζουν μια λύση σε παγκόσμιο επίπεδο διότι καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι καλύτερο για αυτούς από να διατέχουν κίνδυνο διπλής φορολόγησης και πολλαπλασιασμού εθνικών καθεστώτων φορολόγησης. Το αμερικανικό αίτημα όμως καθορίζεται από το γεγονός ότι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του πυλώνα 1 όχι μόνο, που καλείται όχι μόνο ψηφιακές εταιρείε, αλλά και άλλες πολυεθνικές εταιρείε, αυτή η διεύρυνση δημιούργησε αντίδραση από αυτές τις εταιρείε και αυτές οι εταιρείε πιέζουν για να αποφευθεί μια τελική απόφαση, συνοψίζοντας. Νομίζω ότι όσον αφορά τον πυλώνα 1, έχουμε μια καλή τεχνική φύσεως πρόταση, μπορούμε να την επεξεργαστούμε, ούτω ώστε να την εφαρμόσουμε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν καλύτερα τις συνέπειες αυτής της λύσεως για κάθε προπολογισμό, για κάθε κράτος μέλος, αλλά έχουμε ένα τεράστιο ερωτηματικό όσον αφορά την αβεβαιότητα της πολιτικής αποφάσεως. Αυτή η αβεβαιότητα οφείλεται στο ότι η Αμερικανική κυβέρνηση έχει ένα αλλακτικό πρόγραμμα επιλεκτικής φορολόγησης που είναι περίπλοκο σύστημα. Έχουμε προχωρήσει λιγότερο στα άλλα θέματα, στο άλλο θέμα μάλλον, την ελάχιστη φορολόγηση, το ζήτημα αυτό. Βέβαια η κατάσταση είναι λιγότερο επίμαχη όσον αφορά τη σχέση με τη ΣΥΠΑ, θα μας τα εξηγήσει καλύτερα ο διευθυντής του ΟΣΑ που θα μας εξηγήσει καλύτερα τα πράγματα. Ο ΟΣΑ κατάφερε να θεσπίσει αρχές επί των οποίων στηρίζεται η πρόταση που δεν διαφέρουν πολύ από την αρχή που ήδη ισχύει στη ΣΥΠΑ. Εν τη αυτή περίπτωση έχουμε ισχυρή αντίδραση από μικρά κράτη-μέλη, από τη Σιγκαπούρη και από άλλα κράτη-μέλη και ίσως και από μικρές, ε, μάλλον μεγαλύτερες αναδυόμενες οικονομίες. Στον πυλώνα λοιπόν 2 η κατάσταση δεν είναι πιο δύσκολη και πιο επίμαχη, αλλά έχουμε προχωρήσει λιγότερο πλευράς τεχνικής από ότι στον πυλώνα 1. Ε, τελικό σημείο που θέλω να θίξω, μας ανετέθη, ανετέθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ευρωπαϊκές προτάσεις. Να προχωρήσουμε βάσει ευρωπαϊκών προτάσεων αν δεν καταφέρουμε φέτος να συμφωνήσουμε στον πυλώνα 1 και στον πυλώνα 2 ε, στον ψηφιακό τομέα και στην ελάχιστη φορολόγηση. Είναι πολιτικό θέμα, αλλά να καταστήσω σαφές ότι τώρα δεν εξετάζουμε ένα σχέδιο Β, ακόμα και να εξετάζουμε τεχνικής φύσεως λύσεις επικεντρωνόμεθα επί του βασικού προγράμματος, προγράμματος Α, δηλαδή να στηρίξουμε τις λύσεις του ωσα και των G20, διότι η παγκόσμια λύση θα ήταν κάτι πάρα πολύ καλό για την παγκόσμια οικονομία και θα διευκολύνει κατά πολύ και μας. Στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια να θεσπίσουμε αυτή την φορολόγηση αν η λύση αυτή είναι παγκόσμια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε θα δώσω τώρα το λόγο στον Πασκάλ Αρμάν από τον ΩΣΑ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, και καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε. Εγώ θα επικεντρωθώ λιγάκι στον τίτλο του τμήματος αυτού, ότι ξεκινήσαμε το ταξίδι για ένα νέο φορολογικό σύστημα. Ας πάμε λίγο πίσω στο 2008. Είχαμε την χρηματοπιστωτική κρίση που κατέστησε τις κυβερνήσεις, της τράπεζα κοινοβούλια να αντιληφθούν ότι θα έπρεπε να ξεκινήσει κάποια φορολογική ρύθμιση στην παγκοσμιοποίηση. Έχουμε βέβαια φορολογική δικαιοδοσία, αλλά όλοι και οι καταναλωτές και όλοι κατάλαβαν ότι δεν υπήρχε ικανοποιητικός συντονισμός. Έτσι σιγά σιγά προχωρήσαμε πρώτα απ' όλα στη διαφάνεια, να σταματήσει δηλαδή το τραπεζικό απόρριτο και αυτό παντού στον κόσμο, με ελάχιστα σημεία να μην έχουν ακολουθήσει, λίγες χώρες δεν το έχουν κάνει ακόμα, Παναμάς για παράδειγμα, αλλά σιγά σιγά προχωράνε και έπειτα ακριβώ υπήρξε και το θέμα της ε, διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών που προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ψήφισμά σα, το αναφέρατε και νωρίτερα. Ευχαριστώ την Επιτροπή επίση και τον Επίτροπο για τα καλά τους λόγια και άκουσα αυτά που είπατε για σχέδιο Β η δικιά σας η είναι πολύ σημαντική κάθε φορά που κάνουμε ένα παραπάνω βήμα για ένα νέο διεθνές σύστημα. Μπορεί να μην είναι το τελευταίο βήμα, αλλά σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να κάνουμε. Αυτό που διακυδεύεται είναι η ικανότητα των κυβερνήσεων και των δικαιοδοσιών να φορολογήσουν δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα ε, στην επικράτειά τους, η την επιχείρηση βρίσκεται με φυσική παρουσία στην επικράτειά τους ή όχι. Πρόκειται λοιπόν για επιχειρήσεις που έχουν χρήστες, που μπορούν να πουλούν αγαθά, αλλά σήμερα δεν φορολογούνται οπουδήποτε και στη δικαιοδοσία όπου δρούν. Γιατί υπάρχουν ε, κανόνες, κεντρικοί θα λέγαμε, που δεν έχουν προσαρμοστεί στη σημερινή κατάσταση. Και καταλήγουμε μερικές φορές να έχουμε μηδενική φορολόγηση, καθόλου φορολόγηση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να σταματήσει πια αυτή η στρέβλωση που κι εσείς το νιώθετε και σας απογοητεύει η σημερινή κατάσταση γιατί δεν μπορούμε να φορολογήσουμε κάποιες επιχειρήσεις και το φαινόμενο αυτό διωγγώνεται όλο και περισσότερο δεδομένου ότι έχουμε όλο και περισσότερο ψηφιακή οικονομία. Τα τελευταία τρία χρόνια πάντως και από τότε που έκανε την φορολογική της μεταρρύθμιση οι Αμερικοί Ηνωμένε Πολιτείε, δηλαδή που πήγε από το 35% στο 21%, από τότε οι Ηνωμένε Πολιτείε συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις με δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας αναφέρθηκε και νωρίτερα είναι ε, νέα φορολογικά δικαιώματα στις χώρες. Δηλαδή δίνουμε περισσότερα φορολογικά δικαιώματα στην δικαιοδοσία της αγοράς που σημαίνει ότι δικαιούνται να φορολογούν ακόμα και αν δεν υπάρχει φυσική παρουσία μιας επιχείρησης. Δηλαδή πρέπει να βρούμε και να δημιουργήσουμε ένα νέο δίκτυο πωλήσεων και μέρος του κέρδους των επιχειρήσεων να φορολογείται στην δικαιοδοσία όπου ασκούν δραστηριότητες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα το αν ε, έχουν φυσική παρουσία εκεί ή όχι. Και όταν υπάρχει φορολόγηση, υπάρχει σε χαμηλά επίπεδα. Εμείς αυτό που θέλουμε να διασφαλίσουμε είναι ότι ε, τα κέρδη θα φορολογούνται βάσει κάποιου κανόνα, κάποιας εξίσωσης στην ε, δικαιοδοσία όπου ασκούνται και οι εμπορικές δραστηριότητες. Επιπλέον από αυτά τα φορολογικά δικαιώματα ε, θέλουμε να έχουμε και περισσότερη φορολογική βεβαιότητα γιατί οι επιχειρήσεις για να ανθίσουν χρειάζονται ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον, να είναι σίγουρε ότι δεν θα δίπλο φορολογούνται. Δουλεύουμε και πάνω σε αυτό. Ο πυλώνα 2 λοιπόν είναι η δημιουργία ενό ελάχιστου φόρου και το έκανε στη μεταρρύθμιση τη ε, η Αμερική και θέλουμε και εμεί να διασφαλίσουμε ότι μία επιχείρηση εφόσον φορολογείται κάτω από ένα ποσοστό στη χώρα που δραστηριοποιείται, η έδρα της επιχείρησης αυτής μπορεί να αναλάβει την διαφορά και να υποφεληθεί από τη διαφορά ανάμεσα στην ελάχιστη φορολόγηση και την δικιά της. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε όλες οι χώρες να το εφαρμόσουν, να διασφαλίσουν μια ελάχιστη φορολόγηση και αν δεν το κάνει αυτό μια χώρα να φροντίσουν οι υπόλοιπε ε, γι' αυτό. Πριν από μερικές εβδομάδες είχαμε μια ε, συνάντηση με 137 μέλη σε ισότιμη βάση, όλοι εκτό από την Κύπρο είναι μέλη αυτού του Inclusive Framework, όπως το ονομάζουμε, και συμφωνήσαμε για ένα τεχνικό έγγραφο που περιγράφει τον πυλώνα 1, αλλά και κάποια στοιχεία από τον πυλώνα 2 και θα εξετάσουν και οι Υπουργοί Οικονομικών την επόμενη εβδομάδα. Και μετά ερχόμαστε στον Ιούλιο. Πρέπει να έχουμε μια πολιτική συμφωνία η προθεσμία είναι τον Ιούλιο με την επόμενη συνεδρίαση αυτού του πλαισίου, του Inclusive Framework και θα εξετάσουμε την αμερικανική πρόταση που λέει ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται σε θελοντική βάση. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει σε θελοντική βάση φορολόγηση. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ε, ξεκινήσει, θέλουν να προχωρήσουν, αλλά βάζουν κάποιες προϋποθέσεις που για μας είναι δύσκολες. Έχουμε αρκετές εβδομάδες να προχωρήσουμε και σε τεχνικό επίπεδο για να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία. Αυτό διακυδεύεται τώρα. Αν αποτύχουμε, πράγματι δεν υπάρχει σχέδιο Β και το σχέδιο Γ είναι το χάος. Είναι εμπορικό πόλεμος που θα ξεκινήσει αν υπάρχουν ε, φορολογικές διενέξει. Οπότε η πίεση είναι μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε, και πολύ θα χαρούμε αν ξέρουμε ότι έχουμε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο η κυρία Γκρόσδανα Πέριτς. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμοι συναδέλφοι και συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Οι φόροι είναι η κυριότερη και σημαντικότερη πηγή εσόδων κάθε κράτους. Για την άμεση φορολογία αποφασίζει αυτόνομα κάθε χώρα βάσει συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την έμεση φορολογία ε, ενεργεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις πολιτικές της. Τα κράτη-μέλη ασχολούνται κυρίως με την άμεση φορολογία, γιατί είναι απόλυτα στο δικό τους έλεγχο. Και μάλιστα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες η άμεση φορολογία προσφέρει τα περισσότερα κρατικά έσοδα λόγω της ευκολίας συγκέντρωσής τους και των υψηλών φορολογικών συντελεστών που επιβάλλονται. Η άμεση φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ρυθμίζεται άμεσα από τις ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις, αλλά υποφύεται στα κράτη-μέλη να διαμορφώσουν τη φορολογική τους πολιτική και να συλλέξουν του φόρους τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρώνονται άμεση φόροι που προσδιορίζουν και την ανταγωνιστικότητα των κρατών μέλων. Τέτοια άμεση φόροι είναι δύο, ο φόρος εισοδήματο και ο φόρος επί των κερδών. Ο ρόλος του κοινοβουλίων είναι η ε, παροχή συμβουλών σε ό,τι αφορά την ε, άμεση φορολογία ε, και κυρίως η την τήρηση των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια λοιπόν της άμεσης φορολογίας καλό θα ήταν να υπάρχει μία ε, ε, ελάχιστη εναρμόνιση και να αποφευχθεί, να η διπλή φορολόγηση. Σίγουρα ε, η έμεση φορολογία είναι σε μεγάλο βαθμό εναρμονισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ακόμη χώρος και περιθώριο βελτίωσης. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε το σύστημα ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζονται συνθήκες ε, ισότιμου ε, ανταγωνισμού. Θα πρέπει να έχουμε ισχυρή στήριξη για την ε, πλήρη εναρμόνιση του φόρου προστιθέμενης αξίας και διαβουλεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να συνεχίσουμε τις εργασίες και να ολοκληρώσουμε το, την εναρμόνιση του ΦΠΑ. Επίσης, στα πλαίσια της άμεσης φορολόγησης χρειάζεται κάποιο συντονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες οικονομικές προκλήσεις γιατί οι σημερινές φορολογικές διατάξεις ε, αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του 20 του προηγούμενου αιώνα. Έχουν δηλαδή ε, μείνει πια απαρχαιωμένες και ακατάλληλες. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε προσπάθειες ε, για να καταλήξουμε σε πιο δίκαιους, ε, σύγχρονους και αποτελεσματικούς φορολογικούς κανόνες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές προκλήσεις και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Στα πλαίσια της άμεσης φορολογίας, κάθε κράτος μέλος είναι ελεύθερο να ασκήσει την ε, φορολογική του πολιτική που θεωρεί κατάλληλη για τις εθνικές ανάγκες. Υπό τον όρο όμως ότι σέβεται τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι βασικές προτεραιότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η άρση των φορολογικών εμποδίων στην διασυνοριακή οικονομική δραστηριότητα, η καταπολέμηση του αθέμετου φορολογικού ανταγωνισμού και της φοροδιαφυγής και η πρόθεση καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών αρχών σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την καταπολέμηση των φορολογικών απατών. Η εναρμόνιση της φορολογικής πολιτικής στα θέματα της άμεσης φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξυπηρετούσε και την υλοποίηση των ευρύτερων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμού ανάπτυξη με αποτελεσματικό έλεγχο και μείωση της νόμιμης φοροαποφυγής. Επίσης, ε, θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε ενιαίους κοινούς ε, κανόνες για την ενιαία ε, κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση στη φορολογία επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και μείωση του διοικητικού άχθους και για τη διοίκηση αλλά και για τους φορολογούμενους, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την ισότιμη μεταχείριση όλων των φορολογουμένων. Ε, ένα νέο φορολογικό πλαίσιο στα πλαίσια της ψηφιακής οικονομίας που δεν αναγνωρίζει όρια και σύνορα θα εξασφάλιζε καλύτερη ε, αντιμετώπιση των ε, νέων φορολογικών προκλήσεων και κυρίως φορολόγηση των ψηφιακών εταιριών εκεί που δημιουργούν τα κέρδη τους γιατί οι μεμονωμένες φορολογικές εθνικές πολιτικές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις, ε, τους ψηφιακούς κολοσσούς και τις πολυεθνικές που ενεργοποιούνται στο διαδίκτυο. Και μονομερή μέτρα φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας ε, δημιουργούν διαφορετικά φορολογικά συστήματα και απομακρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από μια ενιαία προσέγγιση και μια ενιαία αγορά. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα νέο φορολογικό πλαίσιο για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας και μάλιστα αυτό να γίνει σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για να αποφευθεί η αποδυνάμωση της θέσης των εθνικών κυβερνήσεων και να καλύψουμε το έδαφος και να παρακολουθήσουμε τον ταχύ ρυθμό εξέλιξης των ψηφιακών εταιριών. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Χάνς Μίκελμπαχ. Ευχαριστώ αγαπητέ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα της δίκαιης φορολόγησης των επιχειρήσεων και η απέτηση για μεγαλύτερη διαφάνεια στο φορολογικό τομέα καθώς η καλύτερη καταπολέμηση της φοροαποφυγής και η προώθηση της φορολογικής πολιτικής είναι κάτι που μας απασχολεί επί σειρά ετών στα Εθνικά Κοινοβούλια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όλος ιδιαίτερος στον ΟΣΑ και στο, στη συνόδους των G20. Αφετηρία της προσπάθειας ήταν το πώς ξέφευγαν οι εταιρείες του διαδικτύου από τη φορολόγηση και πολλές εταιρείες που κινούνται σε παγκόσμια κλίμακα. Υπήρχαν και τα προβλήματα των κενών στην εθνική φορολόγηση. Οι χώρες, οι, οι διάφορες εταιρείες εφάρμοζαν φοροαποφυγή. Υπήρχαν συμφωνίε περί φορολογικών σε διάφορα κράτη-μέλη και όλα αυτά οδηγούσαν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, κυρίω για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει που βλάπτονται όλο ιδιαίτερω από αυτέ τι πολιτικέ. Έτσι δε περαιτέρω, θέλαμε να έχουμε ένα σύστημα ΦΠΑ που να προστατεύεται από τις απάτες. Δεν το πετύχαμε αυτό. Πολλά κράτη-μέλη παλεύουν με αυτά τα προβλήματα. Πώς μπορούν να καλύψουν τα κενά που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και στην ψηφιοποίηση της οικονομίας. Υπάρχει γεωγραφική κινητικότητα της φορολογητέας βάση σε μεγάλο βαθμό και μπορούμε να το καταπολεμήσουμε αυτό μόνο σαν μια ενιαία κοινότητα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε να έχουμε μια, ε, έναν κάτωθι αγώνα στον αφορά τη φορολόγηση και ανταγωνισμό. Ε, πρέπει να έχουμε δίκαιους όρους για τον ανταγωνισμό. Αγαπητοί συνάδελφοι, εξυπακούεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΣΑ έχουμε πετύχει πολλά. Το πρόγραμμα των G20 Φερρυπίν για τη διάβρωση του, της, της φορολογητέας βάσεως και τη μετακύληση, μεταφορά των κερδών. Όσον αφορά το BEPS έχουμε πετύχει κάποια πράγματα. Όσον αφορά τη φορολόγηση όμως των ψηφιακών εταιριών, χρειάζεται να επιβληθεί ένας φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και το ίδιο ισχύει και για τα παράγωγα και τις πωλήσει σε μεγάλη κλίμακα και θα πρέπει να υπάρχει και μια δίκαια ενεργειακή φορολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πετύχει λίγα μέχρι τώρα όσον αφορά αυτούς τους τομείς και η κατάσταση που διαμορφώθηκε είναι ατυχής. Κάποια κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει με μονομερή μέτρα και βιαστικά θα έλεγα. Και οι βιαστικές λύσεις ε, είναι επιζήμια για την διεθνή κοινότητα και έγιναν μεταρρυθμίσεις φορολογικές και στις Ηνωμένε Πολιτείε και οδηγηθήκαμε σε αλλαγέ και αλλάξανε και οι θέσεις των, οι διαπραγματευτικές των ΗΠΑ. Υπήρχαν αρχικά ελπίδες, αλλά στη διάσκεψη ασφαλείας του μονάχου που διεξήχθη, είδαμε ότι δηλώθηκε ότι, ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη φορολόγηση στο ψηφιακό τομέα ε, στη ΣΥΠΑ και πρέπει και εμείς να ενωθούμε στην Ευρώπη. Στην, στην Task Force του ΟΣΑ δεν αναφέρεται μια αποτελεσματική βάση φορολόγησης, φορολογική βάση, δεν τονίζεται παρκώς αυτό μιλάει για ανακατανομή της φορολόγησης και των φορολογικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων φορολόγησης. Ακολουθούμε ολιστηρό δρόμο για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ενώσεως και των κρατών μελών. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε μετακίνηση των δικαιωμάτων φορολόγησης προς τα κάτω. Και υπάρχουν και προβλήματα και εμπόδια όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων. Αυτή η προσέγγιση είναι επικίνδυνη για τους εξαγωγείς κυρίως. Λοιπόν, οι εξαγωγές πρέπει να προσεχθούν και θα πληγούν ιδιαίτερα εξαγωγής από την προσέγγιση. Πρέπει να το εξετάσουμε το θέμα. Η Γερμανία είναι ε, συνεισφορέας μεγάλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν χάσει φορολογικά έσοδα, ίσως να μειώσει και τη συνεισφορά τη την οικονομική, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό θα είναι επιζήμιο για την εύρυθμη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να πολλαπλασιαστούν σε διεθνέ επίπεδο οι πρωτοβουλίε επικεντρωνόμενε με μια ελάχιστη φορολογητέ βάση για να αποφυφθεί η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή. 12,5% ε, είναι αυτή η βάση που συζητείται, είναι η βάση των συζητήσεων, όμως πρέπει όλες οι χώρες, πέρα από τα ποσοστά και τα νούμερα, όλες οι χώρες θα πρέπει μετά να είναι σε θέση να παρετηθούν από διορθωτικά και συμπληρωματικά μέτρα που θα εφάρμοζαν, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα dumping φορολογικό. Εμείς και σε επίπεδο ΩΣΑ και G20 θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, να ηγούμεθα για να αντιταχθούμε στη φοροδιαφυγή και στη φοροαποφυγή. Κυρίως να αποφύγουμε να υπάρχει μια διάβρωση της φορολογητέας βάσης. ευχαριστώ. Και περνάμε στη συζήτηση, στην οποία θα προεδρεύσει ο συνάδελφος Μπόρις Λάλοβατς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ ευχαρίστω να προεδρεύσω τη συζήτηση που θα διαρκέσει μισή ώρα. Να σας υπενθυμίσω ότι κάθε ομιλητής θα δικαιούται να μιλήσει δύο λεπτά το πολύ. Ξεκινούμε με τον κύριο Σταύρο Καλογιάννη από τη Βουλή των Ελλήνων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο για την ε, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Σε διοικητικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια οι δράσεις της Ένωσης έχουν ενισχυθεί σημαντικά προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία των φορολογικών αρχών των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης και την ενδυνάμωση της φορολογικής συμμόρφωσης. Σε νομοθετικό επίπεδο είναι σημαντικό να αποτιμηθούν οι φορολογικοί κανόνες και η αποτελεσματικότητά τους, με σκοπό να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που αποτελεί μείζωνα πρόκληση, προσφέρει σημαντικά ωφέλη και ευκαιρίες. Οι ισχύοντες φορολογικοί κανόνες είναι σχεδιασμένοι για επιχειρήσεις με φυσική παρουσία και δεν έχουν προσαρμοστεί απολύτως στην ψηφιακή εποχή, με αποτέλεσμα ψηφιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, με φυσική έδρα σε τρίτη χώρα τεχνολογική κολοσσοί και διαδικτυακές πλατφόρμες να μην φορολογούνται στην Ευρώπη όπου καταγράφονται τα κέρδη τους με δίκαιο τρόπο. Αυτό το γεγονός διαβρώνει τη φορολογική βάση και οδηγεί στην απώλεια πολύ σημαντικών φορολογικών εσόδων. Η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης μιας εταιρείας πρέπει συνεπώς να προσαρμοστεί το συντομότερο, ώστε να περιλαμβάνει και την ψηφιακή δραστηριότητα των εταιριών σε αγορές χωρίς φυσική παρουσία. Η Ελλάδα επιθυμεί τη θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων, προκειμένου οι επιχειρήσεις αυτές να υφίστανται, συγγνώμη, να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία με τον ΟΣΑ είναι θετική. Αναφορικά με τη φορολογία της ενέργειας, οι περιβαλλοντικοί φόροι μπορούν να αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της Ένωσης. Πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Οι ιδιαιτερότητες όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία στηρίζεται στην ακτοπλοεία για τη σύνδεση των νησιών με την υπηρετική χώρα και η όποια επιβολή φόρων στα καύσιμα ναυσιπλοείας θα επιβαρύνει σημαντικά τις ακτοπλοϊκές μεταφορές. Σας ευχαριστώ θερμά. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Επόμενος. Κοκόσοφ, από το Κρατικό Κοινοβούλιο. Αξιότιμοι συμπρόεδροι, αξιότιμοι συναδέλφοι σας και συνάδελφοι. Η ψηφιακή οικονομία αποτελεί ένα νέο παράγοντα ανάπτυξης και γι' αυτό η φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών είναι από τα πιο σημαντικά οικονομικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ψηφιακή πολυεθνικοί κολοσσοί δραστηριοποιούνται παντού στον κόσμο, αλλά προτιμούν να φορολογούνται στις χώρες ε, με χαμηλή, χαμηλό μηδενικό φορολογικό συντελεστή και ουσιαστικά μετατοπίζουν τα κέρδη τους εκεί και αποφεύγουν την ε, φορολόγηση. Κάποιε χώρε έχουν επιβάλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών. όμω η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται ραγδαία, θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειέ μα και να καταλήξουμε σε συνένεση για την φορολόγηση τη ψηφιακή οικονομία, ώστε να μην έχουμε απώλεια φορολογικών εσόδων μερικών κρατών μελών. Είναι περίπλοκο και διεθνέ αυτό το θέμα. Και μόνο διεθνώς θα μπορούσαμε βιώσιμα να, να αντιμετωπίσουμε αυτή την φορολογική πρόκληση και να μειωθεί ο κίνδυνος της διπλής φορολόγησης ε, και να αποφευθεί και απώλεια φορολογικών εσόδων για πολλές χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος, ο κύριος Ζωέλ Ζηρού από τη Γαλλία, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ε, το γνωρίζετε, η Γαλλία έχει εγκρίνει νομοθεσία η οποία είναι και ρεαλιστική και φιλόδοξη όσον αφορά την φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας και λέω ότι είναι ρεαλιστική γιατί εμπνέεται από το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ίδιο θέμα. Συνεπώς είμαστε από τους πρώτους που αναλάβαμε αυτή την πρόκληση και την αντιμετωπίσαμε και λέω ότι πρόκειται για πρόκληση γιατί όντως δύσκολες ήταν πολλές και ακόμα τις βλέπω. Εγώ ήμουν εισηγητής για το κείμενο αυτό και ε, λέγαμε κάθε φορά ότι προσοχή γιατί ο Λευκός Οίκος ε, σας ε, κοιτάει τι κάνετε. Τα ψηφιακά δεν έχουν σύνορα έτσι κι αλλιώς και μια φορολογική πολιτική για να είναι αποτελεσματική πρέπει να έχει και κοινό μέτωπο. Οπότε άκουσα πριν αυτά που είπατε για τις διαπραγματεύσεις στον ΩΣΑ όσον αφορά το σύνολο των διατάξεων και θέλω να γνωρίζω το εξής για τα ψηφιακά ακριβώ. Ποια είναι τα κύρια εμπόδια που εντοπίζετε εσείς και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων γιατί ξέρετε η φορολογία η γαλλική οδήγησε σε μία παύση. Οπότε εγώ θέλω να ξέρω ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να δούμε πότε μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Πιστεύω ότι εφόσον επανεκλεγεί ο πρόεδρος Τραμπ θα επηρεαστεί αυτό το χρονοδιάγραμμα υποθέτω. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Τζεντιλόνη για τις προκαταρτικές του παρατηρήσεις, ιδιαίτερα φιλόδοξες όσον αφορά τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας. Συγκεκριμένα όμως θέλω να ξέρω ποιος είναι ο χάρτης πορείας που ακολουθείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Τανκ Πάρελ, Ευρωβουλευτής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και καλωσορίζω και εγώ εδώ τους συναδέρφους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Πρέπει πιο συχνά να συναντιόμαστε, ιδιαίτερα στο θέμα της φορολόγησης, όπου η πίεση είναι μεγάλη. Πίεση από τους ψηφοφόρους μας που βρίσκουν άδικο, είτε είναι στο εξέτες στην αριστερά, να μην πληρώνουν φόρους οι μεγάλες πολυεθνικές, ενώ αυτοί πληρώνουν. Αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη πίεση που έχουμε από αυτούς. Και η φορολόγηση των επιχειρήσεων είναι πεπαλαιωμένη. Ξεκίνησε από τα μέσα του 20ου αιώνα, τώρα είμαστε στον 21ο. Πρέπει να αλλάξει αυτή ριζικά. Η δεύτερη πίεση είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των χωρών και δεχόμαστε έτσι απειλές από διάφορες χώρες και αποδυναμώνεται η δικιά μας θέση. Πολύ θα θέλαμε, βέβαια, να αλλαξει αυτη ριζικα η δευτερη πιεση ειναι ο ανταγωνισμο μεταξυ των χωρων και δεχομαστε ετσι απειλε απο διαφορες χωρες και αποδυναμωνεται η δικια μα θεση πολυ θα θελαμε βεβαια να δουμε επιτυχια στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, τα και ο Πασκάλ Ντεμόν, να έχουμε πράγματι επιτυχή κατάληξη στις διεθνείς αυτές διαπραγματεύσεις. Και το τονίζω ότι δεν είναι μόνο για τον πυλώνα 2, για την ελάχιστη φορολόγηση, έχει να κάνει και με τον πρώτο πυλώνα, που ουσιαστικά αποτελεί μια ουσιαστική αλλαγή στο φορολογικό σύστημα για να καταλήξουμε σε πιο εξυγχρονισμένους κανόνες φορολόγησης των επιχειρήσεων, όπου επιχειρήσεις θα πληρώνουν φόρο εκεί όπου δραστηριοποιούνται. Πραγματικά. Αυτή η αλλαγή πρέπει να προκύψει. Πάντω, ελπίζω να έχουμε επιτυχεί διαπραγματεύσει. Κοιτάω τον κύριο Τζεντιλόνι εδώ. Επίση, χρειαζόμαστε μια ισχυρή κοινή θέση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση για την φορολόγηση τη ψηφιακή οικονομία έχουν ε, κολλήσει Πρέπει οι Ηνωμένε Πολιτείε να επανέλθουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων και είναι δικιά μα ευθύνη να πετύχουμε και ημών των Ευρωβουλευτών αλλά και των βουλευτών από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Να καταφέρουμε αν μη τι άλλο αυτό. Μην κοιτάτε μόνο τι μπορείτε να κάνετε για τη χώρα σα. κοιτάξτε τι μπορείτε να κάνετε και για την Ευρώπη και τι μπορείτε να κάνετε για να πετύχουμε δίκαια φορολόγηση. Να ψάξουμε λοιπόν να βρούμε νέου τρόπου. Όχι μόνο τελάχιστα δικαιώματα φορολόγησης αλλά και την ελάχιστη φορολόγηση. Ήδη είναι καλό σημείο εκκίνησης αυτό. Σας ευχαριστώ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Μπόζιτσα Μάκαρα από την Κροατία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, το φορολογικό σύστημα της Φορολογικής Ένωσης θα πρέπει να είναι δίκαιο και αποτελεσματικό θα πρέπει να εξασφαλίσει να μην ε, φορολογούνται διπλά τα ίδια έσοδα σε δύο διαφορετικές χώρες μέλη. Και στο μέτρο που υπάρχει τέτοιο πρόβλημα θα πρέπει να διατοπίζουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Με τους νέους κανόνες από την 1η Ιουλίου του 2019 η επίλυση φορολογικών διαφορών έχει απλουστευτεί αρκετά. Τα δικαιώματα των μικρών επιχειρήσεων και των ιδιωτών που έχουν πρόβλημα με τις χρηματικές ουραίες λόγω της διπλής φορολόγησης είναι πολύ περισσότερα πια αλλά θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα αυτό. Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές θα πρέπει να εκδικάζουν τις φορολογικές διαφορές σε εύλογο χρόνο και να απεφεύγονται οπωσδήποτε κολλησιεργίες. Δυστυχώς όμως αυτό στην πράξη συμβαίνει ακόμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Γιάν Κράινερ από την Αυστρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό να εξισορροπήσουμε εκ νέου τα φορολογικά μας συστήματα. Παρόμοια κατάσταση στην Αυστρία, όπως και σε άλλες χώρες. Τη δεκαετία του 70, περίπου 75% του εθνικού εισοδήματος πήγαινε σε εργασία και τα υπόλοιπα πήγαιναν σε ε, κεφάλαιο και πλούτο. 75% των φόρων προήλθαν από εργασία και κατανάλωση και περίπου 25% από κεφάλαιο ε, φορολόγηση εταιρείων και πλούτου. Δίκαιη φορολόγηση. Εν τω μεταξύ, η κατανομή του εθνικού ε, εισοδήματο είναι 60% από εργασία και τα υπόλοιπα από κεφάλαιο και πλούτο. Και η φορολόγηση για κατανάλωση και εργασία 80% και μόνο 20% από κεφάλαια και πλούτο και προσιακά στοιχεία. Αν πάτε σε ένα καφενείο και πάρετε ένα ε, γλυκό και τρώτε ένα 40% του γλυκού και πληρώνετε 20% του λογαριασμού. Αν το κάνετε αυτό θα έχετε προβλήματα μάλλον που, που τρώει 60% και πληρώνει 80% του λογαριασμού. Και την άλλη μέρα θα έχετε πρόβλημα με την αστυνομία. Αυτό δεν ισχύει για την ώρα. Μάλλον θα έχετε πρόβλημα την επιβολή αυτής της νομοθεσίας. Ε, υπάρχει πρόβλημα με τις εταιρείε που πληρώνουν το δίκαιο τίμημα και πρέπει να κάνουμε πολλά. Πρώτα απ' όλα, ελάχιστη φορολόγηση εταιριών. Δεν μπορούν να εφαρμόσουμε αυτό ε, είναι πολύ χαμηλή η φορολόγηση των εταιριών. Πρέπει να αυξηθεί αν θέλουμε να πληρώνουν δίκαιε φορολόγηση εταιρείε. Μετά χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια. Γίνονται τώρα συζητήσεις. Σε τι οφείλονται συζητήσεις. Περισσότεροι άνθρωποι ανακάλυψαν το πόσο λίγα πληρώνει οι μεγάλες εταιρείες. Και χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια. Με τη διαφάνεια βγήκαν αυτές οι πληροφορίες. Μετά θα πρέπει τα, τα τα φορολογικά, τους φορολογικούς παραδείσους και στην Καραϊβική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξαλείψουμε. Το των φόρων των εταιριών που δεν καταβάλλονται στην Αυστρία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες γιατί τα κεφάλαια πάνε κυρίως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, φορολογικούς παραδείσους. Δεν έχω πρόβλημα τη διπλή φορολόγηση. Το πρόβλημα είναι η μηδενική φορολόγηση. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Προς τον κύριο Πασκάλ του ΩΣΑ έχω μια ερώτηση. Μιλήσατε για κάποιο τύπο, κάποια προσέγγιση, μια φόρμουλα αναφέρατε. Ε, τι έχετε υπόψη σας, τι μόρφη θα μπορούσε να έχει αυτή η λύση. Ευχαριστώ. Κυρία Μπίρκιτ Μάλσαχ, Ίνκερμαν, από τη Γερμανία. Καλημέρα, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Έχω ένα πρόβλημα όσον αφορά την ίδια την προσέγγιση που ακολουθείτε. Δηλαδή το πραγματικό πρόβλημα κατά την άποψή μου προέρχεται από τη φορολόγηση των επιχειρήσεων. Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από εκεί, από τη ρίζα, από την έννοια της σταθερής οργάνωσης του συστήματος. Να μην ξεκινάμε οικοδομώντας ένα νέο φόρο διότι οι φόροι, και αυτό ισχύει και για τη φορολογία των εταιριών, πρέπει να καταβάλλονται οι φόροι εκεί που ασκείται η οικονομική δραστηριότητα. Μετά υπάρχει ένα θέμα που αφορά άλλους ιδιωτές στη Γερμανία. Η Γερμανία είναι μια χώρα όπου έχουμε το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο φορολόγησης εν συγκρίση με το Βέλγιο. Αν έπρεπε τώρα να αυξήσουμε ακόμα παραπάνω τους φόρους στη Γερμανία, θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες. Κυρίως εάν σε γενικό παγκόσμιο επίπεδο γίνεται λόγος για ελάχιστο επίπεδο φορολόγησης. Ξέρουμε ότι η φορολόγηση άπτεται της εθνικής κυριαρχίας. Αν θέλουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα λοιπόν, θα πρέπει να βρούμε τα αίτια. Το πρόβλημα δεν είναι ότι είναι πολύ χαμηλοί φόροι που καταβάλλονται και που ζητούνται και απαιτούνται, αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχουμε ανεπαρκή φορολογικά καθεστώτα ξεκινώντας από την φορολόγηση των εταιριών. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε από την έννοια της σταθερής οργάνωσης, να φορολογήσουμε δηλαδή στη βάση. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πολλούς ομιλητές εδώ, μην ε, ζητάτε άλλη ερώτηση παρακαλώ. Η κυρία Φραντσέσκα Ντονάτο, Ευρωβουλευτής, είναι η επόμενη. Ευχαριστώ πολύ. Συζητώντας για Διεθνές Σύστημα Φορολόγησης, πρέπει να επικεντρωθούμε στα εξή. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου, το θέμα της βιωσιμότητας της φορολογίας. Γιατί αν έχουμε ιδιαίτερα υψηλούς φόρους, αυτό μπορεί να έχει ε, κυκλικό ε, αντίκτυπο. Ενώ, αν αντίθετα όπως σε άλλες χώρες, έχουμε ε, dumping φορολογικά συστήματα και αθέμητο ανταγωνισμό, δεν μας συμφέρει. Συνεπώς, η βιωσιμότητα της φορολογίας είναι το πρώτο και μας οδηγεί στο δεύτερο, που έχει να κάνει με τη σύγκληση των συστημάτων φορολόγησης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ελάχιστο φορολογικό επίπεδο, αλλά και ένα ανώτατο επίσης ε, φορολογικό επίπεδο, φορολογικής πίεσης, που δεν θα πρέπει να είναι παραπάνω από το διπλάσιο του ελάχιστου ορίου. Το τρίτο θέμα είναι το θέμα της ανταγωνιστικότητας των ε, παικτών και των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε άλλους που δεν είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πολύ διαφορετικές προδιαγραφές όσον αφορά την παραγωγή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή και τις χώρες εκτός. Ας σκεφτούμε αν μη τι άλλο τους νέους κανόνες που προκύπτουν από τη Νέα Πράσινη Συμφωνία. Συνεπώς, αν δεν υπάρξει επαναεξισορρόπηση και αν δεν εισάγουμε φόρους, ένα πράσινο φόρο ας πούμε, σε αγαθά τα οποία παράγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων απέναντι στις μη ευρωπαϊκές. Και το τελευταίο που χρειάζεται είναι το θέμα της αποτελεσματικότητας της φορολόγησης απέναντι στα κρυπτονομίσματα. Γιατί έχουμε ένα νέο κόσμο, ε, νέο σύστημα πληρωμών. Και αναρωτιέμαι η φορολόγηση πώς μπορεί να είναι αποτελεσματική ελέγχοντας τις κινήσεις αυτές των κρυπτονομισμάτων. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ελένη Σταύρου και από την Κύπρο παρακαλώ. η Κύπρος στάσεται υπέρ της ενίσχυσης της διαφάνειας, του δημοκρατικού ελέγχου και της λογοδοσίας σε φορολογικά ζητήματα. Η εντατικοποίηση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και της διοικητικής συνεργασίας ανάμεσα στις φορολογικές αρχές των κρατών μελών είναι καθοριστική σημασίας για τη διασφάλιση μιας δίκαιης και αποτελεσματικής ενιαίας αγοράς, καθώς και για την πάταξη των φαινομένων της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Τα φαινόμενα αυτά είναι διασυνοριακά και δεν μπορούν να επιληθούν αποτελεσματικά μονομερώς, καθώς η αντιμετώπιση τους απαιτεί συλλογικές προσπάθειες, συντονισμό και συνέργειες ανάμεσα στις εθνικές, φορολογικές αρχές. Η αναγκαιότητα άμεσης καταπολέμησης των πιο πάνω φαινομένων διαπιστώνεται αν αναλογιστούμε πόσο επιζήμια είναι τα φαινόμενα αυτά για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, δεδομένου ότι οδηγούν στην απώλεια σημαντικών φορολογικών εσόδων που θα χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση δημοσίων πολιτικών, παραδείγματο χάρη την παροχή δωρεάν εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη. Η φορολόγηση συνιστά ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτει η κυβέρνηση τη κάθε χώρα για χάραξη τη κοινωνική και οικονομική τη πολιτική αποδοκιμάζουμε την προωθούμενη κοινή βάση φορολόγησης εταιριών και την ενδεχόμενη εναρμόνιση των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών διότι εκτιμούμε ότι θα είναι επιβλαβή για την κυπριακή οικονομία πιστεύουμε ότι η φορολόγηση θα πρέπει να παραμείνει στη δικαιοδοσία των κρατών μελών ως αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα. η κύπρος είναι απομονωμένη αγορά μικρού μεγέθους χωρίς χερσαία διασύνδεση σε μια σταθή περιοχή με μεγάλες εξωτερικές προκλήσεις. τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της κυπριακής οικονομίας είναι περιορισμένα και ο χαμηλός φορολογικός συντελεστής είναι κέρια σημασίας για την προσέλκυση επενδύσεων και τη διατήρηση της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας ποιότητας της κυπριακής οικονομίας. Σας ευχαριστούμε. Okay. Thank you. Σας ευχαριστώ. Ο Κρίστοφ Τοζεύσκη από την Πολωνία είναι ο επόμενος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η οικονομία σίγουρα έχει αλλάξει ε, δυναμικά λόγω και της ψηφιοποίησης. Εξού και η ανάγκη Φορολόγηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων των μεγάλων ψηφιακών πολυεθνικών. Στα πλαίσια του ΩΣΑ ε, έχουμε κάποιους φόβους για την πρόταση του ε, πυλώνα 2 σε ό,τι αφορά το υποτιθέμενο εισόδημα ή το εικαζόμενο εισόδημα. Πιστεύουμε ότι έτσι ίσως ε, εξουδετερωθούν ε, οι φορολογικές ελαφρύνσεις ε, κάποιων νομικών προσώπων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη ε, ιδιαίτερα στις δραστηριότητες των οικονομικών ζωνών. Θεωρούμε ότι η, ο αποκλεισμό των, των ε, κερδών και τις πραγματικές δραστηριότητες θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Μόνο έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί αν η ιδέα του εικαζόμενου φόρου ε, είναι συμβατή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κάποιες εξαιρέσεις αποκλεισμού. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του πρώτου πυλώνα, ε, ενώ το σημείο α είναι αξιόλογο και θα πρέπει να εξεταστεί. Παρ' όλα αυτά, για, τις, για το φορολογικό συντελεστή Β ή Γ δεν υπάρχουν αρκετές μελέτες ως τώρα, ώστε να στοιχειοδετούν την ε, βασιμότητα αυτών των προτάσεων. Ο κύριος Ερικ Ποκέ από τη Γαλλία, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω την πρωτοβουλία που αναλάβατε για να συμπεριλάβετε και αυτή τη συζήτηση στο πρόγραμμα της συνεδρίασης. Γιατί θα πρέπει συνεχώς ε, να μιλούμε για αυτό το θέμα, όχι μόνο στα πλαίσια του Κοινοβουλίου ή της κυβέρνησης και της δημόσιου διαλόγου, αλλά συνεχώς γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα που οδηγεί σε τεράστιες ε, απώλειες φορολογικών εσόδων στην φορολογία ενός λόγω της φοροδιαφυγής. Υπάρχει ένα δημοσιονομικό λοιπόν ε, ζήτημα και πρόκληση, αλλά και δημοκρατικό ζήτημα. Γιατί αμφισβητεί την ικανότητα των κρατών να εφαρμόσουν τη φορολογική νομοθεσία σε όλους τους φορολογούμενους. Μερικές φορές τα μηνύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αντιφατικά. Ο νέος επιτροπός, ο Thierry Μπρετόν, στις 20 Ιανουαρίου μίλησε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και είπε ότι αν ο ΩΣΑ δεν καταφέρει να συμφωνήσει για φορολόγηση της ε, ψηφιακής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλάβει τις ευθύνε και θα εφαρμόσει τέτοια ψηφιακή φορολογία. Και ενώ τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση ενημερώνει κατάλογο, το, τη μαύρη λίστα των φορολογικών παραδείσων και περιέλαβε τον Παναμά και τις Ιχέλες, αλλά δεν αναφέρει ε, τις Παρθένες νήσους, ε, τις Μπαχάμες, τις Ιχέλες. Γιατί? Γιατί είναι σαφές ότι έχουν διασυνδέσεις με το σύντη του Λονδίνου και το, μετά το Brexit το Ηνωμένο Βασίλειο φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαφύγει των κανόνων και της φορολογικής διαφάνειας. Ποια είναι λοιπόν η πραγματική βούληση Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς ε, έχει κατάσταση ό,τι αφορά τη βούληση των κρατών μελών, των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ μιας νομοθεσίας των ψηφιακών δραστηριοτήτων, γιατί υπάρχουν ενδιασμοί, είχαμε μια παλινδρόμηση στον πιεριτ πέρυσι, ε, είχαμε και τον Νοέμβριο κάποια προβλήματα, πώς έχει κατάσταση στα κράτη-μέλη και θα μπορούσαμε ίσως επι, επιτέλους για τα φορολογικά ζητήματα να καταργήσουμε τον κανόνα της ομοφωνίας και να περάσουμε σε μια ειδική πλειοψηφία στις ψηφοφορίες. Ο κύριος Γιάννης Κόποτσεφ έχει τώρα το λόγο από την Τσεχία. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα από την πλευρά μου να μιλήσω για την κοινή φορολογική βάση, κάτι το οποίο αναφέρθηκε πολλές φορές μέχρι τώρα. Το θέμα αυτό δεν είναι βέβαια νέο. Ε, συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετά χρόνια. Και δεν πρόκειται απλώς για μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Είναι επίση και ένα από τα βήματα που κάνουμε για την φορολογική εναρμόνιση. Πολλοί αναφέρθηκαν στην φορολογική εναρμόνιση, αλλά εγώ θέλω να σας πω να προσέξετε, γιατί η φορολογική εναρμόνιση περιορίζει το φορολογικό ανταγωνισμό. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι η φορολογική εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε αύξηση του φορολογικού βάρους των ε, φορολογούμενων, δηλαδή τόσο τους Ευρωπαίους πολίτες όσο και τις επιχειρήσεις. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι η υψηλή φόρη σημαίνει αδυναμία στην ε, οικονομική μεγένθηση και η φόρη που είναι υψηλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο είναι και μία από τις αιτίε για την οποία έχουμε τόσο πολύ αδύναμη ανάπτυξη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Ξέρω ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την φοροαποφυγή, ότι θέλουμε να έχουμε ανταλλαγή δεδομένων για τα φορολογικά δεδομένα δηλαδή, αλλά προσοχή στον ανταγωνισμό που είναι πολύ σημαντικός. Το φορολογικό άκθος δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Και τέλος, ο φορολογικό ανταγωνισμός πρέπει να προστατευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από χώρες με διαφορετικές οικονομικές ε, επιδόσεις ή ορίμανσης. Και δεν έχει νόημα οι πλούσιες χώρες να έχουν το ίδιο φορολογικό βάρος όσο και οι φτωχές, οι οποίες προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Ευχαριστούμε. χαμάκι Φιλανδία τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε. Θα ήθελα από τη δικιά μου τη πλευρά να αναφερθώ στο εξή. Έχουμε εδώ τις σωστές ερωτήσεις, μιλάμε για το σωστό πρόβλημα, γιατί το κύριο πρόβλημα στην ουσία είναι ότι πολύ κεφάλαιο διαρρέει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε από Facebook είτε από άλλες πλατφόρμες που έχουν κέρδη εδώ, όπως η Google, η Amazon και τα λοιπά. Όμως, αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι όταν πληρώνουμε τις επιχειρήσεις αυτές, είτε με τη Visa είτε με την Amex, επίσης έχουν ε, κέρδη. Το βράδυ κοιτάμε το Netflix. Τα κέρδη πάνε στις Ηνωμένε Πολιτείε. Στην πραγματικότητα όμως είναι πάρα πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Το βασικό πρόβλημα που βλέπω εγώ είναι ότι μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων εδώ στην Ευρώπη δίνει κέρδα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, ναι, πρέπει να πετύχουμε ώστε ο χρήστης που χρησιμοποιεί μια υπηρεσία, ο ίδιος ο χρήστης χρησιμοποιώντας την υπηρεσία αυτή να δημιουργεί εκεί που την χρησιμοποιεί κέρδος, φορολογικό κέρδος. Γιατί η χώρα στην οποία προσφέρεται υπηρεσία επίσης πρέπει να έχει έσοδα από την υπηρεσία αυτή. Βέβαια, όλα αυτά θα οδηγήσουν σε τεράστιο διοικητικό άχθος, που θα ήταν και αυτό προβληματικό. Οπότε στην πράξη το πιο εύκολο, κατά τη γνώμη μου, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει η ίδια ε, τέτοιες ψηφικές υπηρεσίες ώστε να αποφεύγεται η διαρροή αυτή κερδών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλιώς να πετύχουμε μια παγκόσμια συμφωνία με τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε. Ιταλία τώρα. Ο κ. Ντανιέρε Πέσκο από την Ιταλία. Θέλω να πω ότι πιθανότατα πρέπει να σεβαστούμε την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφορά το σεβασμό μεταξύ χωρών. Πολλές χώρες κάνουν φορολογικό ντάμπινγκ έναντι άλλων χωρών και υπόκειται σαν ειδικά αποτελέσματα. Λέμε ότι είμαστε δημοκρατικοί, θα πρέπει να βρούμε μια λύση δημοκρατική λοιπόν, ούτως ώστε αυτό το φορολογικό ντάμπινγκ να μην γίνεται πια. Όσον αφορά το τελευταίο θέμα του, φορολο... του web taxing, η Ιταλία όπως η Γαλλία και η Αυστρία θέσπισε ένα φορολο... φορολόγηση στο διαδίκτυο και θα ήταν καλό και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να το κάνουν, ώστε να μπορούν να αντιταχθούν με σοβαρό και αποφασιστικό τρόπο έναντι ενδεχομένων αντιπίνων από οικονομικές δυνάμεις όπως είναι η ΕΠΑ. Πάντως, όσον αφορά το web tax, να δώσω μια συμβουλή σε όλους. Εμείς έχουμε ξεπεράσει κάπως τους ορισμούς του ΩΣΑ ήδη εδώ και αρκετά χρόνια. Παραδείγματο χάρη, έχουμε δει ότι μια επιχείρηση από το εξωτερικό που έχει μια ε, δράση σε μια χώρα και έχει συνεχή παρουσία οικονομική στην επικράτεια της χώρας αυτής δημιουργείται έτσι ούτως ώστε να μην έχει, βλέπουμε ότι δεν έχει φυσική παρουσία στην επικράτεια. Μια εταιρεία μέσω πλατφόρμα web μπορεί να δραστηριοποιείται, που βρίσκεται σε άλλη χώρα, αλλά βγάζει κέρδο στη χώρα, θα πρέπει να πληρώνει φόρου σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, τα καταφέραμε μέσω των ορισμού του πώ διοργανώνεται η εταιρεία. Παρακαλώ, αν μπορείτε, θα μπορείτε να το δείτε αυτό σαν λύση που έχουμε βρει εμεί. Ευχαριστώ. Τώρα στον Επίτροπο να δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και δεν είναι καθόλου εύκολο να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Θα περιοριστώ σε δύο-τρία σχόλια και οι υπόλοιποι συνάδελφοι ίσως θα συμπληρώσουν. Καταρχάς, Έχουμε σημειώσει πολλά επιτέγματα τα τελευταία χρόνια. Και εγώ δεν διεκδικώ τίποτα από αυτά γιατί είμαι νέο μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θεωρώ ότι και όσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαδικασία του ΜΠΕΠ, της διάβρωσης φορολογικής βάσης ε, και της μετατόπισης κερδών, ε, σημείωσαν μεγάλη πρόοδο σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της φορολογικής συνεργασίας, στην καταπολέμηση της φοροαποφυγής και ούτω καθεξής. Βέβαια γνωρίζουμε ότι οι προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας είναι πολλές και μεγάλες. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο κώδικας συμπεριφοράς, ο οδοντολογικός κώδικας και, ε, και το έργο που γίνεται στα πλαίσια της σύνταξης μαύρης λίστας είναι πολύ θετικά. Και θεωρώ ότι και άλλες χώρες όντως θα μπορούσαν, οι άλλες δικαιοδοσίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτό το κατάλογο. Πάντως ε, κάνω μια πολύ ακριβή ανάλυση και δέχομαι ότι θα μπορούσαμε ίσως να βελτιώσουμε τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού. Μάλιστα, κάποια κράτη-μέλη ζητούν να εφαρμόσουμε τέτοιο έλεγχο και στα κράτη-μέλη. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή την πρόταση την υπέβαλε η δανεική κυβέρνηση. Και η απάντησή μου ήταν ότι καταρχήν δεν έχω, πρόβλημα, αλλά θα πρέπει να συντονίσω αυτό το θέμα με τη συζήτηση για ένα παγκόσμιο κατώτατο φόρο γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένα σε αυτές οι δύο διαδικασίες και αν δεν υπάρχει συντονισμός θα δημιουργηθούν προβλήματα. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια κοινή θέση, τι έχει αποφασίσει. Ναι, έχουμε κοινή θέση. Έχουμε καταλήξει κοινή θέση εν ώψη των συζητήσεων που θα γίνουν στον ΟΣΑ το επόμενο Σαββατοκύριακο στο Ριάντ. Και η βάση αυτής της κοινή θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συνεργασία για να βρούμε μια παγκόσμια λύση και για το δεύτερο πυλώνα αλλά και για τον πρώτο πυλώνα. Και δεν ήταν καθόλου εύκολο να καταλήξουμε σε αυτή την κοινή θέση. Και γνωρίζετε κάλλιστα ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Γιατί οι ευρωπαϊκές συνθήκες που δεν τις αλλάζουμε είναι υπέρ της ιδέας ότι οι αποφάσεις για τα φορολογικά θέματα θα πρέπει να λαμβάνονται με ομοφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και τη ρήτρα Πασαρέλα που προβλέπει ομόφωνη απόφαση ε, για την κατάργηση της ομοφωνίας ή για την ε, παρέκκληση από την ομοφωνία. Ούτε και αυτό είναι εύκολο. Οπότε η πολιτική βούληση είναι ξεκάθαρη και δεδηλωμένη, αλλά δυστυχώς ε, δεν έχουμε πάντα αποτελέσματα παρά την πολιτική βούληση που έχουμε. Και υπάρχει το πρόβλημα με τη ρήτρα της ομοφωνίας. Πριν από δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποβάλει πρόταση ακριβώς για την ψηφιακή φορολόγηση και η πρόταση αυτή να βάγισε, δεν υιοθετήθηκε λόγω του βέτου, λόγω της αντίθεσης τριών χωρών μελών. Αλλά αυτοί είναι οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να τους αποδεχτούμε. Και αν δεν θέλουμε να λάβουμε υπόψη άλλες πιθανότητες, άλλες δυνατότητες που μας δίνει το άρθρο 116 για παράδειγμα, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που θα γίνει στο μέλλον. Πολιτική βούληση λοιπόν υπάρχει, υπάρχει και ενότητα, γιατί όπως σας είπα σήμερα το πρωί υιοθετήσαμε μια δήλωση που δίνει σε μένα και στον ε, Κροάτη Υπουργό Οικονομικών που εκπροσωπεί ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ΡΙΑΤ ε, ως ασκών την Προεδρία. Έχουμε λοιπόν εντολή να στηρίξουμε αναφαδό την πρόταση του ΟΣΑ. Και μάλιστα και το G20 προσπαθεί να κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον και να αξιοποιήσει την όθηση που έχει δημιουργηθεί πέρα αυτής της πρότασης. Τέλος, για το φιλοπορίαση τον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα θέματα αυτά. Ε, εγώ στην επιστολή ανάθεσης ε, καθηκόντων μου έλαβα και συγκεκριμένες εντολές για τον οδικό χάρτη. Είναι σαφής λοιπόν ο οδικός χάρτης. Θα πρέπει όμως να καταλήξουμε σε συμφωνία σε διεθνές επίπεδο. Αυτή είναι η αποστολή μου. Αν δεν καταλήξουμε σε παγκόσμια συμφωνία το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση για ρυθμίση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2020 δεν είναι μία ημερομηνία που επιλέξαμε μόνο τυπολατρικά. Γιατί η εθνική νομοθεσία, όχι μόνο η γαλλική, αλλά και η ιταλική και η αυστριακή, η τσεχική αντίστοιχη νομοθεσία και από ό,τι κατάλαβα και η ισπανική νομοθεσία που αποφασίστηκε σήμερα από την ισπανική κυβέρνηση, όλες αυτές οι νομοθετικές προτάσεις των χωρών μελών έχουν την ιδέα Τη ίσπραξη εσόδων από το 2021 λόγω του ψηφιακού φόρου. Αυτό αποφάσισε πρόσφατα και η γαλλική κυβέρνηση και ήδη έχει περιληφθεί στις εθνικές ε, νομοθεσίες των χωρών που σας ανέφερα. Εξού και η κρίσιμη προθεσμία του 2020, ειδικά μετά τις ε, γαλλικές αποφάσεις ε, και ε, δεδομένων των χαρακτηριστικών της γαλλικής νομοθεσίας ε, δεν θα έχουμε έσοδα από τους ψηφιακούς αυτούς φόρους ε, ούτε στα κράτη-μέλη που έχουν θεσπίσει τέτοια ψηφιακά, τέτοιες νομοθετικές διατάξεις. Αλλά το 2021 η κατάσταση θα αλλάξει. Για φέτος δεν θα υπάρξουν αλλαγές. Οπότε θέλουμε παγκόσμια συμφωνία κατά τη διάρκεια του 2020. Και ο δικός χάρτης προβλέπει ότι αν δεν καταφέρουμε να συνάψουμε διεθνή συμφωνία φέτος, θα πρέπει να υποβάλουμε μια ευρωπαϊκή πρόταση. Πάντως, η σύναψη συμφωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο έχει στρατηγική σημασία για μας για να αποφύγουμε εμπορικούς πολέμους και άλλες δυσκολίες και για να θα σπίσουμε ένα νέο διεθνές φορολογικό σύστημα. Κάτι τέτοιο είναι απολύτως απαραίτητο και εξαιρετικά σημαντικό για το μέλλον των οικονομιών μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ. Επειδή δεν έχουμε χρόνο θα είμαι σύντομο. Ποια είναι τα εμπόδια προκειμένου να καταλήξουμε σε κάποια λύση. Υπάρχουν πολλά. Δηλαδή, Πρώτα απ' όλα, νέο σχεδιασμός του διεθνούς φορολογικού πλαισίου. Αυτό βέβαια δυσκολεύει κάπως τις χώρες, αισθάνονται άβολα, γιατί όντω υπάρχουν πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Πρώτα απ' όλα, ε, να δούμε την πρόταση των ΗΠΑ, μετά να δούμε την ισορροπία που πρέπει να πετύχουμε ανάμεσα στα δικαιώματα φορολόγησης και την φορολογική βεβαιότητα για τι αναδυόμενες οικονομίες, για παράδειγμα. Και τρίτον, να λάβουμε υπόψη μα και τι ιδιαίτερότητε κάποιων χωρών. Κάποιες ασιατικέ οικονομίες λένε ότι ε, μπορούν να υποφεληθούν περισσότερο κάποιε ξένες επιχειρήσει από ό,τι άλλες και άρα μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη επιστροφή. Έπειτα πρέπει να δούμε όντως την περίπτωση της ψηφιακής οικονομίας με τις τεχνικές προκλήσεις για τις οποίες πρέπει εμείς να έχουμε κάποιες λύσεις μακροπρόθεσμα, που να κρατήσουν δηλαδή. Μέχρι τον Ιούλιο πρέπει να έχουμε κάτι. Θα έχουμε, δεν ξέρουμε. Εδώ λοιπόν είναι η μεγάλη δυσκολία. Ε, το χρονοδιάγραμμα, η επόμενη συνεδρίαση θα είναι πρώτη και δεύτερη Ιουλίου στο Βερολίνο του πλαισίου. Και πρέπει να έχουμε ήδη κάποια λύση να προτείνουμε προκειμένου αυτή να εφαρμοστεί. Και εννοείται ότι πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα αναπτυχθεί αυτή η νομοθεσία. Με ένα πολυμερές πλαίσιο θα πάρει κάποιο χρόνο. Αλλά πάντως τον Νοέμβριο οι G20 θα πρέπει να έχουν την συμφωνία όλων και γι' αυτό λέμε ότι τον Ιούλιο θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί όλα αυτά. Τώρα αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Μπορεί να χρειαστούν κάποιοι μήνες παραπάνω για την εφαρμογή αυτή καθεαυτή, αλλά πάντως όλα τα στοιχεία της πολιτικής ε, πρότασης για λύση πρέπει να έχουν συμφωνηθεί μέχρι τότε. Και αν θέλετε να δείτε την ρύθμιση που προβλέπουμε, την φόρμουλα, την εξίσωση που προβλέπουμε, να πάτε στο στην ιστοσελίδα μας. Και εκεί θα βρείτε το τόσο της εκατό ε, και πόσο θα είναι στις ιδιαίτερα κερδοφόρες επιχειρήσεις που θα πάρουν ένα κομμάτι. Για να καταλήξουμε δηλαδή σε ένα αναλογικό σύστημα βάση κερδών. Ευχαριστούμε. Ποιος? Κύριος κύριος Μίχελμπαχ θα ήθελα για μία ακόμη φορά να στραφώ προς τη συζήτηση που διεξήχθη. Δεν θέλω να εμποδίσω τον φορολογικό ανταγωνισμό όπως είπε κάποιος. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε ο ποσοστό φορολόγησης. Εγώ μιλούσα για ελάχιστη φορολόγηση. Όταν υπάρχει διαφάνεια, μπορεί τότε να προσφέρονται και κίνητρα για τις επιχειρήσεις. Αλλά αυτό που στο κάτω-κάτω μετράει περισσότερο από όλα είναι η διαφάνεια και πάνω απ' όλα να αποφεύγεται το φορολογικό dumping. Έχουμε μεγάλη διαφυγή εσόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φορολογικών εσόδων και φεύγουν αυτά τα έσοδα και πάνε εκτός επικρατής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το σταματήσουμε, να το εμποδίσουμε, διότι είναι τεράστιο έλλειμμα αυτό που δημιουργείται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλη απώλεια, αυτή η ε, διαφυγή του φορολογικού εσόδου και έχει αντίκτυπο στους πολίτες μας. Και δεν μπορούμε αυτή την ευθύνη να την, να αφήσουμε έτσι, να περάσει έτσι. Διότι δεν έχουμε τον αναγκαίο φορολογικό μηχανισμό για να το αντιμετωπίσουμε. Το να καθορίσουμε ελάχιστο επίπεδο φορολόγησης σε επίπεδο ΩΣΑ στα 12,5% ή λίγο πιο κάτω, τουλάχιστον αν γίνει αυτό, θα έχουμε μια εγγύηση διαφάνειας. Είναι βασικό ζήτημα και πρέπει να παραμείνει βασικό ζήτημα το θέμα του δικαιώματος που έχει κάθε χώρα να επιβάλλει μια φορολόγηση όσον αφορά έσοδα που γίνονται σε μια άλλη χώρα εάν αυτή η φορολόγηση δεν έχει γίνει βάσει μιας ενός ελάχιστου φορολογικού συντελεστή. για να εμποδίσουμε μία ε, μη φορολόγηση. Ο εξυγχρονισμός των φορολογικών μηχανισμών είναι σημαντική πτυχή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν περιπλοκότατα συστήματα φορολογικά. Η Γαλλία και η Γερμανία δημιούργησαν δύο επιτροπές στα πλαίσια των Υπουργείων Οικονομικών ούτω ώστε να εξετάσουν κοινά μέτρα, ε, κοινή προσέγγιση όσον αφορά την φορολόγηση των εταιριών. Είναι μια πρώτη προσέγγιση που θα πρέπει κατά την άποψή μου να καλύψει τελικά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να είναι περιορισμένο πείραμα που αφορά μόνο τη Γαλλία και τη Γερμανία. Όλα τα θέματα αυτά, όπως και το δικαίωμα και η φορολογική ουδετερότητα που ίσως είναι κάτι απαραίτητο για τον εξυγχρονισμό των φορολογικών συστημάτων, όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από πλευράς των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων. Πρέπει να βρούμε λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Κυρία Πέριτς. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω ότι θα βρούμε την καλύτερη λύση για να έχουμε ένα αρμονισμένο σύστημα ΦΠΑ και να συμφωνήσουμε και για κάποιες κοινέ γραμμές για το φόρο εισοδήματος, ώστε να μην επιβαρύνουμε υπερβολικά ούτε τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε τις ε, κυβερνήσεις ή τις χώρες μέλη. Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ επικοδομητική συζήτηση γιατί υπάρχουν πολλές προτάσεις από τα κράτη-μέλη και όλες αυτές οι προτάσεις θα συμβάλλουν στη, στη δημιουργία ενός ποιοτικού πλαισίου ώστε να συνεχίσει να ασκεί ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά και να αναπτύσσεται με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ωραία. Έχουμε καθυστερήσει μισή ώρα. Οπότε έχουμε 20-25 λεπτά μόνο για το δεύτερο τμήμα. Οπότε προτείνω το εξή. Να μην έχουμε εισαγωγικέ παρατηρήσει, να κερδίσουμε έτσι 3-4 λεπτά και να έχουμε 10 παρεμβάσει μονόλεπτε όμως από τους βουλευτέ. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έγκαιρα. Το δεύτερο θέμα λοιπόν είναι από τη διαφάνεια στη βιωσιμότητα. Ε, στόχοι περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομικής διακυβέρνησης. Α, συγγνώμη, βιάστηκα. Ωραία, εγώ θα ξεκινήσω και θα αλλάξουν οι ομιλητές εδώ ε, στο, στο βήμα δίπλα μου. Πρέπει να φύγουν οι προηγούμενοι και να έρθουν οι καινούριοι. Οπότε, επειδή έχουμε χάσει χρόνο, την εισαγωγική μου παρουσίαση θα την κάνω συγχρόνω όσο αλλάζουν θέσεις οι ομιλητές. Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να πετύχουμε τους στόχους του 2030 που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι, πρέπει να καλύψουμε ένα επενδυτικό κενό το οποίο υπολογίζεται σε 180 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε αυτό το στόχο χρησιμοποιώντας και ιδιωτικά και δημόσια κονδύλια. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε εργαστεί για να δημιουργήσουμε το σωστό πλαίσιο ώστε να επαναπροσανατολίσουμε τα κονδύλια προς τη βιώσιμη χρηματοδότηση για να στηρίξουμε την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ε, τη διαφάνεια μακροπρόθεσμα και να δημιουργήσουμε και μια κυκλική οικονομία χωρίς άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή στη συζήτηση αυτή και πέρυσι οι συνομοθέτες κατέληξαν σε δύο νομοθετικές πράξεις. Η πρώτη για τα κριτήρια χαμηλού άνθρακα και η δεύτερη είχε να κάνει με τις απαιτήσει γνωστοποίησης των χρηματοδοτικών υπηρεσιών. Επίσης, έχουμε και την πρότασή μας για την ταξινομία, η οποία ολοκληρώνεται όπου να είναι, που αποτελεί ένα πολύ σημαντικό νομοθετικό στοιχείο. Σήμερα είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και για τα δύο άλλα στοιχεία που είναι η κοινωνική πτυχή και η πτυχή της διακυβέρνησης. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η συνοχή, οι αμοιβέ κτλ. Πιστεύω ότι όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε στη συζήτηση και θα δώσω τώρα το λόγο πρώτα στον Τζον Μπέρικαν που είναι υπηρεσιακός γενικός διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Φύσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε δύο λεπτά, τρία λεπτά κύριε Πρόεδρε. Ah, Θα πω τα μισά, γιατί ήδη καλύφθηκαν αρκετά. Τι θέλω να πω. Να υπενθυμίσω καταρχάς ότι δεν μιλάμε πλέον για τους στόχους ε, της χιλιετίας ευρωπαϊκούς, αλλά ανήκουμε στη Νέα Πράσινη Συμφωνία πλέον. Αυτό το πράσινο σύμφωνο τι κάνει. Βγάζει τη βιώσιμη χρηματοδότηση που ξεκίνησε σαν ένα περιθωριακό προϊόν και έγινε βασική δραστηριότητα της αγοράς και μπαίνει ένα καινούριο πλαίσιο. Τώρα έχουμε στόχο το 2050 να είμαστε ουδέτεροι από πλευρά άνθρακα. Όλοι λοιπόν θα πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους. Τι κάναμε μέχρι τώρα όπως υπογραμμίσατε. Στη δράση για την ε, βιώσιμη χρηματοδότηση, σχέδιο δράση 1, έχουμε τρία νομοθετήματα. Βαθμολόγηση, αποκάλυψη, έλεγχος και η ταξινόμηση. Τι κάνουνε αυτά τα τρία στοιχεία. Βοηθούν τους επενδυτές, επιτρέπουν στους επενδυτές να εντοπίσουν τι είναι πράσινο. Αυτή είναι η ταξινομία, τους δίνει τη γλώσσα. Η αποκάλυψη τους δίνει τις πληροφορίες απαραίτητες να ξέρουν ότι να επενδύουν σε κάτι σε τι επενδύουν και ότι αυτό στο οποίο επενδύουν είναι πράσινο προϊόν και ο κανονισμό περί βαθμολόγηση του δίνει εργαλεία επί των οποίων μπορούν να βασιστούν για να βαθμολογήσουν την απόδοση τη επενδύσεω. Άρα είναι βολικό πλαίσιο. Μία στρατηγική που βοηθά τους επενδυτές να επιλέξουν. Του δίνουμε τα εργαλεία και επιλέγουν για την πράσινη προσέγγιση. Βέβαια, μπαίνουμε σε μια άλλη φάση τώρα, όπω είπα. Ανήκουμε στην πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκή και Έχουμε χρονοδιάγραμμα. Στη νέα διευθέτηση, στη νέα στρατηγική που θα υποβληθεί φέτο. θα μετακινηθούμε από πιο παθητική προσέγγιση σε πιο ενεργητική προσέγγιση. Πρέπει να το κάνουμε αυτό, διότι τώρα έχουμε πλέον 30 χρόνια για να πετύχουμε τα αποτελέσματα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε μέσω περισσότερων κινήτρων για αυτά που πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορώ πω τώρα τι θέλουμε να περιλάβουμε στο πρόγραμμα. Πρέπει να γίνουν δημόσιες διαβουλεύσεις, αλλά έχουμε ιδέες πριν ξεκινήσουμε διαβουλεύσεις σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιες από τις ιδέες θα συμπεριλαμβάνουν περισσότερη δουλειά όσον αφορά την αποκάλυψη στοιχείων, πιο πολύ υποχρεωτική αποκάλυψη στοιχείων και ευρύτερο πεδίο να καλύπτεται. Περισσότερες εταιρείες, κυρίως στο μη χρηματοδοτικό τομέα, διότι ο κανονισμός τώρα εστιάζεται κυρίω επί του χρηματοδοτικού τομέα, ανακαλύπτουν εταιρείε εκτό του χρηματοδοτικού, ευρύτερο πλαίσιο και υποχρεωτική υποχρέωση αποκάλυψη. Περισσότερα στοιχεία να παρουσιάσουν στην αγορά, περισσότερα στοιχεία που απαιτούνται, ώστε οι επενδυτέ να μπορούν να κατανοήσουν τι είναι πράσινο και πώ μπορούν να είναι πράσινε επενδύσει. Θέλουμε να διευκολύσουμε τι επενδύσει σε πράσινα μέτρα καλύτερη τικητοθεσία, καλύτερη χρήση προτύπων και προδιαγραφών, κυρίω ε, ε, το, το πράσινο ομόλογο πρέπει να προχωρήσουμε για να μοχλέψουμε καλύτερα τη δράση του ιδιωτικού τομέα όσον αφορά τις επενδύσεις που θα κάνουν διότι ο δημόσιο τομέα δεν μπορεί μόνο στο να κινηθεί όσον αφορά τη χρηματοδότηση, χρειάζεται και η βοήθεια του ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να κατανοήσουμε επίση ότι ο δημόσιο τομέα επίση θα πρέπει να παίξει το ρόλο του, όχι τόσο αφορά τα ε, δημοσιονομικά, όσον αφορά την πολιτική. Τα εργαλεία που θεσπίζουμε για το ειδικό τομέα, κυρίω η ταξινόμηση αυτή, θα πρέπει να αποτελέσει βάση για δημόσια πολιτική και μέτρα που θα θεσπιστούν, ούτως ώστε να κινηθούμε προς το στόχο του 2050, του στόχους του 2050. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πάει ακόμα στους... δεν αλλάξαμε όσον αφορά την περιβαλλοντική κοινωνική διακυβέρνηση. Λοιπόν, Έχουμε πει ήδη ότι πρέπει να κάνουμε μια κίνηση προς τα εκεί. Δεν θα πρέπει τελειώτης να είναι εχθρό του καλού. Ξεκινήσαμε με το περιβάλλον, με κάποια στοιχεία περί περιβάλλοντος και θα επεκταθούμε. Μετά από αυτό όμως θα πρέπει το θεματολόγιο να κινηθεί σε θέματα διακυβέρνησης και κοινωνικά θέματα που βέβαια θα είναι πιο δυσχερή ζητήματα διότι βασίζονται λιγότερο επί επιστημών αλλά είναι βάση κρίσεως και νομοθεσίας. Αυτή είναι η δέσμευση που αναλάβαμε και έτσι θα κινηθούμε. Θα σταματήσω εκεί και ελπίζω να κάλυψα όλα στα τρία λεπτά που είχα στη διάθεσή μου. Μάλιστα. Και τώρα, τώρα να δώσω το λόγο στον Μπόρις Λάλοβατς. Σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσω κουρατικά. Στην έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2018 αναφέρεται η Γενική Στρατηγική Βιώσιμων Χρηματοοικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκεί αναφέρεται ότι η βιομηχανική επανά... χρηματοδότηση θα πρέπει να έχει δύο άξονες, τη βελτίωση της της βιώσιμης χρηματοδότησης προκειμένου να λαμβάνει υπόψη κριτήρια κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ε, σωστής διακυβέρνησης που θα πρέπει να διέπουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Έτσι, με την σωστή βιώσιμη χρηματοδότηση θα προωθείται η κοινωνικά υπεύθυνη οικονομία που θα εξασφαλίζει ποιότητα ζωής και πλήρη απασχόληση. Είναι λοιπόν ε, σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ε, τη σημασία των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πτυχών και τους συναφείς κινδύνους κατά την κατά τις επενδυτικές μας αποφάσεις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα και να λάβουμε υπόψη ότι για, την, για τις επενδύσεις δεν είναι απαραίτητη μόνο η κερδοφορία ως κριτήριο, αλλά οι επενδυτές ενδιαφέρονται και για τις επιπτώσεις συγκεκριμένων επενδύσεων στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στη διακυβέρνηση. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τέτοια βιώσιμα βιοοικονομικά, λαμβάνοντας υπόψη και αυτά τα τρία χαρακτηριστικά. Μάλιστα, οι εμπλεκόμενοι παράγοντε ενδιαφέρονται περισσότερο για τη δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών των επιχειρήσεων. Και σίγουρα τα περιβαλλοντικά και ελληνικά κριτήρια ε, θέλουν να ξέρουν οι επενδυτέ αν λαμβάνονται υπόψη για την υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων. Έτσι ε, θα αυξηθεί και η απασχόληση αλλά και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επενδυτών στις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Κολτζάνα Πέριτς για να συντονίσει τις ερωταπαντήσεις. Ένας έχει ζητήσει το λόγο, αλλά να σας υπενθυμίσω προηγουμένως ότι η συζήτηση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να συνεχιστεί και αύριο σε 9.30 στην Ολομέλεια. Ε, σας ευχαριστώ. Έχουμε, όπως είπε και η Συμπρόεδρος, ένα μονομιλητή. Ζήτησε το λόγο ο εκπρόσωπος της Πολωνικής Βουλής με ένα όνομα που είναι δύσκολο για προφορά. Ο κύριος Τχουζεύσκι. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε προϋποθέτουν όχι μόνο χρηματοοικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πολύ εύρωστη εσωτερική οικονομική διαχείριση. Για την ενεργειακή και την ψηφιακή μετάβαση χρειάζονται τεράστια οικονομικά κονδύλια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα κράτη-μέλη. Η Πολωνία τα τελευταία χρόνια έχει αντιμετωπίσει όλο και περισσότερες προκλήσεις ε, ε, λόγω της, ε, των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και της αδυναμίας φορολογίας τέτοιων διασυνοριακών οικονομικών δραστηριοτήτων. Χρειάζεται ενίσχυση της συνεργασίας των φορολογικών αρχών και ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Γι' αυτό και η Πολωνία υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες που στόχο έχουν την αύξηση της φορολογικής διαφάνειας και κυρίως ε, την ενίσχυση της ε, ανταλλαγής των πληροφοριών μεταξύ των εφοριών. Εμείς ε, έχουμε τέτοια εμπειρία από συνεργασία με φορολογικές αρχές των κρατών μελών και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων εφοριών και μάλιστα έχουμε προσυπογράψει την σύμβαση για την διοικητική συνεργασία στα φορολογικά θέματα. Είμαστε υπέρ της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και υποστηρίξαμε αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 27 χωρών και των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης, οι δράσεις που έχουμε πραγματοποιήσει έχουν οδηγήσει ένα περιορισμό της φοροαποφυγής και άρα αύξη των φορολογικών μας εσόδων. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι Οι δράσει που αναλάβαμε ε, είχαν ε, την υποστήριξη και της κοινωνίας των πολιτών και μάλιστα προωθήσαμε και ένα πρόγραμμα για, την, ε, για τις κεφαλαϊκές ροές που λαμβάνουν υπόψη και περιφαλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Και μάλιστα η πιο μακροπρόθεσμη προοπτική είναι κάτι που μας προβληματίζει ιδιαίτερος. Μόνο έτσι θα εξασφαλίσουμε ε, αηφόρο χρηματοδότηση και καλύτερη ε, διακυβέρνηση των επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τζον Μπέργεν. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να πω ότι συμφωνώ για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει ένα ρόλο, αλλά δεν είναι και ο μόνος παίκτη. Έχουμε την Πράσινη Συμφωνία και στην Πράσινη Συμφωνία, στα πλαίσια της, θα φροντίσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς μέσω του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, του Invest Europe, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κλπ. κλπ. για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Αλλά συμφωνώ ότι και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να αναλυθούν βήματα. Πρέπει να ε, βοηθήσουν και οι χώρες όσο γίνεται περισσότερο. Και το θέμα της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής επίσης πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά να επικεντρωθούμε για να αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις βιωσιμότητας, που είναι και εθνικές προκλήσεις. Όμως παρόλα αυτά ξέρουμε όταν πρόκειται κυρίως για το κλίμα, αλλά όχι μόνο και για τα κοινωνικά και για τη διακυβέρνηση, δεν θα μπορεί καμία χώρα από μόνη της να τα αντιμετωπίσει και σίγουρα κανένας δημόσιος τομέας. Γι' αυτό και χρειάζονται ιδιωτικά κονδύλια. Και έτσι και η δικιά μου υπηρεσία, ε, το δικό μου τμήμα, αλλά και όλοι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να καταρτήσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα επιτρέψει στον ιδιωτικό τομέα να παίξει το δικό του ρόλο στα πλαίσια όλων αυτών των αλλαγών και προκειμένου να πετύχουμε την βιωσιμότητα. Ευχαριστώ τελευταίος ο κύριος Λάλοβατς. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Είναι όντως πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και θα συνεχίσει να μας απασχολεί και στο μέλλον. Είναι ένα θέμα που αφορά και τη φορολόγηση και την ενία κεφαλαία αγορά και την ε, ανάγκη να ενημερώνονται οι, οι επενδυτές για το κατά πόσο οι επενδύσεις ε, θα επηρεάσουν το περιβάλλον. Και αυτό σε συνδυασμό με τη Νέα Πράσινη Συμφωνία μας υποχρεώνει να εξετάσουμε όλα αυτά. Νομίζω όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινείται στη σωστή πορεία γιατί προσπαθεί αφενός να προωθήσει κάποια φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα και αφετέρου να εξασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια για τους επενδυτές ε, που πραγματοποιούν τις επενδύσεις και θέλουν να ξέρουν αν τα χρήματά τους ε, θα χρηματοδοτήσουν φιλοπεριβαλλοντικά προγράμματα και σχέδια. Σας ευχαριστώ, λέει κυρία Πέρις. Ε, μπορούμε να κηρύξουμε το πέρας αυτής της διακοινοβουλευτικής συνεδρίας Επιτροπής ΕΚΟΝ και να σας καλέσουμε σε ένα κοινό δείπνο που θα παραθέσει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο, προ, ο κύριος David, David ε, σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Κρατικής Βουλής, τον κύριο Γιαντροκόβιτς. Ε, το δείπνο θα παρατεθεί στον οίκο της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Σας ευχαριστώ και συνέχεια στο δείπνο.